να ξεκινήσουμε. Bene, buongiorno a tutti. Καλημέρα σας. Ξεκινάμε. Έχουμε μια ολόκληρη μέρα ψηφοφοριών. Ας ε, καθίσουμε στις θέσεις μας. Ξεκινάμε με την ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Για τεχνικούς λόγους η σημερινή διερμηνία δεν υπάρχει σε όλες τις γλώσσες της Επιτροπής μας. Λείπουν τα φιλανδικά, τα λιθουανικά και τα σλοβενικά. Να σας πω ότι όλη η σημερινή συνεδρίαση μεταδίδεται μέσω web stream στο διαδίκτυο. Και πολλοί θα μας παρακολουθούν. Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών της συνεδριάσης 11 Οκτωβρίου 2012, 5η και 6 Νοεμβρίου 2012, 26 Νοεμβρίου 2012. Αγαπητοί συνάδελφοι, πάμε τώρα στην ψηφοφορία μας όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής λάβαμε, όπως θα γνωρίζετε, χιλιάδες ε, τροπολογίες, περίπου 8.000 τροπολογίες. Οι εισηγητές μας εργάστηκαν πολύ σκληρά, μαζί με όλους τους σκιώδεις εισηγητές, για να εξευρεθούν συμβιβασμοί στα σημαντικότερα ζητήματα που προτείνονται. Πριν ε, ξεκινήσουμε, να κάνω κάποιες εισαγωγικές ε, παρατηρήσεις, οι οποίες ισχύουν για τις άμεσες πληρωμές και που θα επαναληφθούν και για κάθε ένα από τα τέσσερα χαρτοφυλάκια τα οποία, στα οποία θα ψηφίσουμε σήμερα και αύριο. Συνάδελφοι, δεν θα ψηφίσουμε επί των εκθέσεων για πρώτη ανάγνωση, αλλά επί προτάσεων για διαπραγματευτική εντολή. Σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 2 και 70α του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος μας είναι να ψηφίσουμε τη διαπραγματευτική εντολή ε, στην Ολομέλεια του Μαρτίου 2013. Εντολή θα παρτίζεται από προτάσεις τροποποίησεων των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εφόσον όπως γνωρίζουμε η πρικοδότηση οικονομική που σχετίζεται με τις νομοθετικές προτάσεις είναι απλώς ενδεικτική η εντολή θα μπορούσε να καθοριστεί τελικά και οριστικά μόνο όταν θα επιτευχθεί μια συμφωνία επί της προτάσεως του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Η διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 70 μας επιτρέπει να προχωρήσουμε τις διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση κοινή γεωργικής πολιτικής και εν απουσία ενός πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου, ήτι, για να είμαι ακριβή η Επιτροπή μας επιφυλάσσεται του ελέγχου του χαρτοφυλακίου αυτού και μπορεί να καθορίσει τώρα την προσωρινή της θέση χωρίς να γνωρίζει το ακριβές διαθέσιμο ποσό για τη χρηματοδότηση κοινή γεωργική πολιτική, αλλά ελπίζουμε βέβαια να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο αμέσω μετά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια που προβλέπεται για την σύνοδο του επομένου Μαρτίου. Επιτρέψτε μου να επενθυμίσω ότι λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού των τροπολογιών δεν είναι πάντα εφικτό να εγγυηθούμε το 100% της συνοχής όλου του κειμένου μόνο με, την, με το κατάλογο των ψηφοφοριών. Αν υπάρξουν αντιφάσεις στο κείμενο μετά, το, μετά την ψηφοφορία, η γραμματεία θα πρέπει να κάνει τις δέουσες προσαρμογές, κυρίως όσον αφορά τις τελογικές σκέψεις, που θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν βεβαίως το περιεχόμενο των άρθρων. Αν υπάρχει αμφιβολία θα ψηφίσουμε, θα κάνουμε μια ψηφοφορία παραπάνω για να εγγυηθούμε το στο επίπεδο δημοκρατίας στην ψηφοφορία. Αν όλοι οι συμβιβασμοί, προσοχή, για όλες τις συμβαστικές τροπολογίες, οι ψηφοφορίες θα γίνουν με ηλεκτρονικό τρόπο. Όπως η ηλεκτρονική θα είναι και η πρώτη ψηφοφορία που θα λάβει η χώρα τώρα όσον αφορά την τροπολογία Reimers, την αρχική, και ηλεκτρονική, ηλεκτρονικές θα είναι οι ψηφοφορίες όσον αφορά το capping. Στα υπόλοιπα σημεία θα προσπαθήσουμε διανατάσσως τη χειρός να ψηφίσουμε για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Καλώς. Θα ήθελα συνάδελφοι να ανακοινώσω σε όλους ότι δεν θα δεχτώ προφορικές τροπολογίες αν υπάρξουν προφορικέ τροπολογίες, αν υπήρχαν προφορικέ τροπολογίες θα είχαμε σοβαρά χρονικά προβλήματα. Αρκετοί συνάδελφοι μου ζήτησαν να κάνω αυτή τη διευκρίνηση και γι' αυτό σα παρακαλώ, επειδή έχουμε δύο πολύ σημαντικέ μέρε, σα παρακαλώ λέγω να βοηθήσουμε ένα τον άλλον για να κάνουμε καλή δουλειά. Πριν ξεκινήσουμε τώρα με τι ψηφοφορίε και πριν κάνουμε μια δοκιμή όσον αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών καρτών και των ψηφοφοριών, θα ήθελα να ρωτήσω αν ο Λουίς θέλει να πάρει το λόγο ε, για να μιλήσει για λίγο. Λουίς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα μακρηγορήσω γιατί έχουμε πάρα πολύ δουλειά μπροστά μας. Αλλά πριν την ψηφοφορία ήθελα απλώς ε, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την ηλεκτρονική του συνεργασία, τους βοηθούς τους, την γραμματεία της Επιτροπής Γεωργίας, τις γραμματείες των πολιτικών ομάδων. Ξέρω ότι είναι ε, μία δουλειά που αλληλοσυνδέεται με όλους και έτσι κατορθώσαμε να φτάσουμε αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Σμποβέ. Ήθελα να πάρω το λόγο σε σχέση με το άρθρο 70. Αυτό μου θέτει ένα πρόβλημα κατανόησης. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι κάτι καινούριο, καθώς ε, υιοθετήθηκε το Νοέμβριο και επομένως ε, για αυτή την καινούργια διαδικασία αναρωτιέμαι με τον τρόπο που θα το κείμενο στην Ολομέλεια. Αν κατάλαβα το άρθρο 70 προσδιορίζει το πλαίσιο διαπραγματεύσεω τη Κομισιόν ε, στον τριμερή διάλογο. Αυτό δεν μου θέτει πρόβλημα, όμω αυτό που μου δημιουργεί πρόβλημα είναι ότι σήμερα θα ψηφίσουμε. Πολύ ωραία. Το κείμενο θα διαβαστεί στην διάσκεψη των Προέδρων. Πολύ ωραία η ψηφοφορία θα γίνει ε, στην Ολομέλεια, στις τροπολογίες που μπορεί να παρουσιαστούν ε, από τις ομάδες ως εναλλακτικέ ε, της Επιτροπής. Αν κατάλαβα καλά, αυτό σημαίνει ότι δεν θα συζητήσουμε για το σύνολο του κειμένου για να μπορούμε να τη βελτιώσουμε, να το τροποποιήσουμε στην Ολομέλεια. Έτσι λοιπόν ε, θα βρεθούμε με το κείμενο που θα έχει ψηφιστεί σήμερα, που δεν είναι σχεδόν οριστικό, και αν υπάρξει τροποποίηση στην ολομέλεια βάσει τροπολόγιων που θα έχουν κατατεθεί από τι ομάδε. Αυτό μου θέτει σοβαρό πρόβλημα για τη δημοκρατική διαδικασία και για το ότι η Ολομέλεια θα αναγκαστεί να μπορεί να κάνει μια βάθος συζήτηση ε, επί του κειμένου. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Δηλαδή, εγώ θα καταψηφίσω την πρόταση αυτή, εκτό και να μου δώσετε κάποια εξήγηση που να μπορέσει να με πείσει και να κατανοήσω τα πράγματα. Πρόεδρο, καταρχήν, θα ήθελα να καθησυχάσω τον κύριο Μποβέ. Έχουμε μια πλήρη συζήτηση στην Ολομέλη. Δεν υπάρχουν ε, αμφιβολίες ερμηνευτικέ για το άρθρο 70. Θα έλεγα λοιπόν να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα με την ψηφοφορία. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε με ένα τεστ για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Να ψηφίσουμε για την Επιτροπή μας. Λοιπόν, δοκιμή. Ποιος είναι υπέρ της Επιτροπής Γεωργίας. Però, abbiamo una larga maggioranza. Έχουμε βρει επιλοψηφία. Attenzione, il gruppo SD c'è un voto di... Λοιπόν, για τους σοσιαλιστές ε, υπάρχει μια ψήφος παραπάνω. Μπορείτε να κάνετε έναν έλεγχο. Allora, cancelliamo e facciamo un'altra voto, ok? Un'altra? Allora, un altro voto di prova. Λοιπόν, άλλη μια δοκιμή. Ποιος είναι υπέρ της Επιτροπής μας. Παρακαλώ, ψηφίζουμε. Είναι εντάξει, μάλιστα, ωραία. Επομένω, ε, είμαστε προσεκτικοί, μην αλλάξετε κάτι, γιατί τώρα είναι όλα εντάξει. Να ξεκινήσουμε με την τροπολογία Reimers, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ποιο είναι υπέρ τη τροπολογία 111. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 11 ψήφι υπέρ. Ας περάσουμε στους συμβιβασμούς. Συμβασμός α υπέρ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Είστε το όλο. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το συμβασμό Β. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συνδεσμός C, γάμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στο συνδεσμό C, α. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται και ο ΣΥΑ. Περνάμε στο συμβασμό D, δέλτα. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας για το συμβασμό D. Εγκρίνεται. Περνάμε σε δύο επιλογές για το greening. Περνάμε στην επιλογή 1 του συνδεσμού ε, ή άρχεται η αρχεται Πέρασε. Εγκρίνεται. 22-21. Και τώρα να περάσουμε στο F. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε το συνδεσμό G. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ωραία. Συνεχίζουμε. Με ανάταση χειρός. Περνάμε στροπολογία 325. Υπέρ ποιος είναι. Για την 325. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 327, 326, 327 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. 328 Χόσλινγκ υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Πάμε στον 332 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 3.43 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 344 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 345 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται να ψηφίσουμε τον έλεγχο του προπλησμού 8 υπέρ κατά εποχές πρέπει να κάνουμε έναν έλεγχο ηλεκτρονικό, άρχεται η ψηφοφορία για το 8. Πέρας, απορρίπτεται. Να περάσουμε στο 2. 356. Υπέρ, ανάταση κατά. Εποχές, απορρίπτεται. Λοιπόν, 9. Ένα του προπολογισμού υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 3. Ρέτζι 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύε 4. Υπέρ. Κατά. Κάνουμε ένα έλεγχο. Άρχεται η ψηφορία για την TV4. Πέρασε. Απορρίπτεται. Άρθρο 4, 358, Γκίρλινγκ, υπέρ. Κατά. Εποχές, απορρίπτεται. 359, υπέρ. Κατά. Εποχές, απορρίπτεται. 360 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 361 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 362 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 363 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 364 υπέρ κατά εποχέ απορρίπτεται 365 υπέρ κατά εποχέ απορρίπτεται η 20 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 366 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται υπέρ υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται υπέρ υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται υπέρ υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 3-1 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται Envy 11 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 373 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 374 υπέρ κατά εποχές να ελέγξουμε το 374 του κ. Νταντάν. Άρχεται η ψηφορία. Σωστατόλη. όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 378. Πάμε στο 378. Νταντάν υπέρ. Κατά. Εποχές. Πάλι έλεγχο για το 378. Δεν ήταν και λυπή. Άρχεται η ψηφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται για μία ψήφο. 384. Ηλεκτρονική ψηφορία. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 383. Ντότς, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 386 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 387 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 388 υπέρ κατά εποχές θα έλεγα ότι απορρίπτεται 381 Νίκολσον υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 3,82 82 όσλινγκ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 380 Νικολέσκου υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ένβη 11 υπέρ. Κατά. εποχέ απορρίπτεται. Κόντ 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 389 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 390 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 391 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται NV12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πάμε στο 394 υπέρ όχι 408 όσλινγκ υπέρ. Κατά. εποχέ απορρίπτεται. Έρευ 14. 409 υπέρ κατά. Εποχές απορρίπτεται. 410. παρήρα και λοιπή υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 411 γιατί υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται 412 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πάμε 455 όσοι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 456 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συγγνώμη. 456 εγκρίνεται. 459 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 460 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23 το συγγητή υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 461 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 463 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 464 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 465 υπέρ. Κατά αποχές θα λέγαμε γκρίνεται. 466 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 469 περ κατά αποχές απορρίπτεται 470 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 471 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 473 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 474 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για το 474. Ψήφισε το όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 475. Υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 476 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 477 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 478 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 εισήτης, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 481 Κατά. εποχές απορρίπτεται. 482 υπέρ. Κατά. εποχές απορρίπτεται. 1.17 υπέρ. Κατά. εποχές απορρίπτεται. 484 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. 484 link. Πέρας απορρίπτεται με ευρία πλειοψηφία. 485 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 486 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άνβη 17 υπέρ κατά εποχέ, απορρίπτεται. 489 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στο 493 υπέρ. Όχι. Συγγνώμη. Κύριε πρόεδρο. Λοιπόν, για το Λεμπρούν. 496 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 497. 497 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 499 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 500 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο για το 500. Έχουμε βρει πλειοψηφία να ελέγξουμε αυτό ζητάτε. Άρχεται η ψηφορία για το 500. Πέρας. Απορρίπτεται. Συνεχίζουμε με ένα τεσχυρό. 502. Υπέρ. Κατά. εποχέ Απορρίπτεται. 503. Υπέρ. Κατά. Εποχέ. Απορρίπτεται. 504. Υπέρ. Κατά. Εποχέ. Απορρίπτεται. 505 υπέρ κατά εποχές απορρίπτει Πάμε στο άρθρο 7. 508, υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 513 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 516 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 525. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 527. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 526. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 528. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 529 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 530. 531 διορθώνει ο πρόεδρος υπέρ. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 533 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 534. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα έλεγα γκρίνεται. Να ελέγξουμε. Για τον 538 Ρας Γκαρσία. Συγγνώμη, 534 Ρας Γκαρσία και λοιπή. Άρχεται ψηφορία. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται. Άρθρο 8. 535. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 536. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. 2.695 υπέρ. Κατά. Εποχές. Θέλω ότι εγκρίνεται. Να κάνουμε έναν έλεγχο για το 2295. Γκάβριλ Νικολέσκου, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεν να δούμε. Απορρίπτεται. 28. Μετασχυρός. Υπέρ. Κατά. Τυχές, εγκρίνεται. Λοιπόν, να πάμε τώρα στη τροπολογία 685 του άρθρου 10 με τα υπέρ. 685 υπέρ κατά. Αποχές απορριπτωται 686 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 687 υπέρ κατά σε απορρίπτεται. 688 υπέρ κατά Πιστεύω απορρίπτεται. Για το 688 Σιλβέστρης έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 689. Άρχεται η υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 690. Νίκολσον υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 691 Όσλινγκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 692 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 694 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6,95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6,97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6,99 Γκάμπριελ υπέρ κατά αποχές θα να γκρίνεται έλεγχος για το 6,99 άρχεται η Πέρας. Απορρίπτεται. Λοιπόν, 2.296 για repair. Κατά. Αποχές. έλεγχος. 2.296. Άρχεται ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ισοπαλία. Είχαμε και μία εποχή. Μάλιστα. Προχωράμε. Άρθρο 11. Για το κάπινγκ, τα μετατόρια. Υπέρ, ε, ποιος είναι υπέρ για το 700. Για το μπλοκ αλφα, Μπλοκ αλφα υπέρ. Κατά. Εποχές. Και λίγο απορρίπτεται. Πάμε στο μπλοκ β. Προσοχή. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Block C. Υπέρ. Κατά. εποχές, Απορρίπτεται. Block D. Υπέρ. Κατά. εποχές, Απορρίπτεται. Block E. Υπέρ. Κατά. εποχές, Απορρίπτεται. <coughs> Θέλετε να γίνει έλεγχος για το ε. Για το E. Ελέγχουμε. Πέρας. το βρέως. Μπλοκ F. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. G. Υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. Block H. Υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. Block I. Πρέπει να έχουμε ετοιματική ψηφοφορία. Ξεκινάμε. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 754 υπέρ. Όχι. 37. Ψηφίζουμε 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Περνάμε στο Globe J υπέρ. Μια στιγμή. Yeah, until 6769. Possiamo votare? Λοιπόν, Block J. Έχουμε τις πρώτες πέντε τροπολογίες. Υπέρ. Κατά. Αποχές υπορρίπτεται. Συνεχίζουμε με τα μεμονωμένα άρθρα. 769 Lion. Υπέρ. Κατά. Να κάνουμε έλεγχο. Άρχεται ψηφορία για το 769. Πέρας. Έλεγα εγκρίνεται. Όχι, απορρίπτεται. 767 ρόντους του. Υπέρ. Αυτά. Αποχές και δεν είναι δύσκολο. Πρέπει να κάνουμε έναν έλεγχο για το 767. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. 767 και απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε την 38. Υπέρ του άρθρου 38 του εισηγητού. Κατά. Εγκρίνεται. 774. Όσλινγκ υπέρ. 774. Κατά. Απορρίπτεται. 776. Σκοτάκια άλλη υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 775 υπέρ κατά εγκρίνεται μάλλον. Ας γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 775 μακίνες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 777 λεγιάρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 779 και στον υπέρ. Κατά. Άποχες. Θα έλεγα ότι εγκρίνεται. Έλεγχος. 779 Κόστιγκζερ, ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας και απορρίπτεται με ισοπαλία. 780 Φερέιρα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 782 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 778 Α, συγγνώμη, 784 Νίκολσον υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 791 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 792 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 793 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία για την 793 793 πέρας και Απορρίπτεται και εδώ μισοψηφία. 789 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 794 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 801 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συγγνώμη. Έλεγχος για την 801. Γκάμπριλ. Άρχεται η ψηφοφορία. 801. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 796 υπέρ. 796. Κατά. Εγκρίνεται. 797 υπέρ. Α, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. Πάμε στο άρθρο 12. 803 υπέρ. 803 κατά αποχές απορρίπτεται. 804 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ε, κάνουμε μεγάλο άλμα. Άθρα 870. Στο 870 τρόπο λέει. 870 μακίνες. Υπέρ. 870 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 869 downtown υπέρ 869 κατά αποχές έλεγχος θα κάνουμε έλεγχο για την 869 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. απορρίπτεται. 44 υπέρ, διανατάσσεως της χειρός υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 871, 871 υπέρ, κατά, θα έλεγα ότι απορρίπτεται αλλά σε ελέγξουμε. 871 Γκάμπριελ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας.

2297 ψηφισατόρι απορρίπτεται. 873 υπέρ. 873 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Πάμε στο άρθρο 17. 874 Νίκολσον υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 875 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 876 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Άλλο μεγάλο άλμα, συνάδελφοι. Molto bene. Stiamo procedendo bene. va... Πολύ καλά πάμε. Αν πηγαίνω πολύ γρήγορα πείτε το μου. 1214. Νίκολσον. Συγγνώμη. 1215. 1215. 1215 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1219 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος προπολογισμού 17 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 12-17 Νίκολσον υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 12-18 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 12-20 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 12-21 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 12.23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θα έλεγα. Έλεγχος 12.23 τελάως άρχεται η ψηφοφορία έλεγχος ηλεκτρονικός. 12.23 έλεγχος ψηφίσατε όλοι απορρίπτεται. 12.24 υπέρ 12-24 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12-25 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12-27 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12-28 λούλινγκ υπέρ, κατά, υπέρ, συγγνώμη, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Όχι, 1228 Λούλινγκ ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι για τη 1228. Πέρας. Απορρίπτεται. 1229 Σμιθ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1230. 1230 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1231. 1231 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12.32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12.33 υπέρ, κατά, αποχές, θα έλεγα ότι εγκρίνεται. 12.33 θα γίνει έλεγχος. 12.33 έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. 12.33. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. 12.34 Σμιτ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12.38 Μαγκίνες υπέρ, 12.38 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται θα έλεγα. 12.39 υπέρ, κατά, αποχές, θα έλεγα ότι απορρίπτεται, όμω πρέπει να γίνει έλεγχο, Ζητώ συγγνώμη. 1239 Γκάμπριελ, έλεγχο. 1239 ψηφίσατε όλοι. Πέρα ψηφοφορία για το 1239 και απορρίπτεται. 62 υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά, κατά, εγκρίνεται. 1242 υπέρ, κατά, απόχέ, απορρίπτεται. Και άλλο μεγάλο άλμα, αγαπητοί συνάδελφοι. Μόλτο μπένε. Είστε έτοιμοι. Says a Non diciamo le pagine che sono diverse. E allora Άρθρο, μάλλον τροπολογία 1863, Νίκολσον. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται θα έλεγα. Συνεχίζουμε, 1865, Γιάρ και άλλοι, υπέρ, κατά, Αποχές. Θα έλεγα ότι απορρίπτεται. 1800 έλεγχος. Καλώς. 1865. Ας κάνουμε έναν έλεγχο. Γιάρ και άλλοι. Λοιπόν, ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. Και προσοχή. Εγκρίνεται. Δίκιο είχατε. Μπράβο, Γιάρ. 1867. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1868. 1868 υπέρ. Όχι. Πάμε στο άθρο 4. 1869 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1871 Νίκολσον υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1872. Αντρίο και άλλοι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος, όχι έλεγχος. 1874 υπέρ. 1874 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1875 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1876 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1877 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται μάλλον. Να κάνουμε έλεγχο. 1877 ten, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικός έλεγχος. 1877 πέρας ψηφοφορίας για την 1877 η οποία απορρίπτεται. Πάμε στην 1878 Αντρίου υπέρ, της 1878 υπέρ, κατά, απορρίπτεται θα έλεγα. Ψηφίζουμε την NV29, NV29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1879, 1879 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1880 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1881 Μισό λεπτό. Ψηφίζουμε τη 1882, λέει ο Πρόεδρος. 1882 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1884. 1885 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1886 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 1887 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 1888 Ντόρφμαν υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 1888 έλεγχος. Ντόρφμαν 1888 ηλεκτρονικός έλεγχος. πέρας ψηφοφορίας και απορρίπτεται. 18 18-89 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 18.90 ταραμπέλα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 18.91 πατράων έβες υπέρ, κατά, απορρίπτεται μάλλον. 18.92 υπέρ, 18.92 Ντόρφμαν υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 1893 Λεχιάρικ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. MV30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1894 Ντόρφμαν υπέρ κατά κατά αποχές απορρίπτεται. 1895 υπέρ 1894 έλεγχο. Εντάξει, 1894 Ντόρφμαν Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. 1894. Να απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Πάμε στη 1895. 1895. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα έλεγα ότι απορρίπτεται και αυτή. Με την ίδια διαφορά. 1897. Άρθρο 35-1898. Γιάρ και άλλοι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1900. Ντόρφμαν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, συγγνώμη. Έλεγχος για τη 1900. Ντόρφμαν. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται. Σωστά. 1901 ταραμπέλα. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Και εδώ. 1901. Ψηφίσατε για τη 1901 ταραμπέλα. Πέρας. Απορρίπτεται και αυτή. Ψηφίζουμε τη 1903. Μάγερ. 1903 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. και άλλα αλματάκια θα κάνουμε. Ψηφίζουμε την Καρόνα 2003 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2004 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2005 απορρίπτεται συγγνώμη απορρίπτεται απορρίπτεται 2005 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2006 με την ίδια διαφορά. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 2007. Όλοι κατά. Άρθρο 38. Ξεκινάμε. Μισό λεπτό. Ξεκινάμε με τη 2009. Υπέρ. 2009. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2011 υπέρ κατά αποχές έλεγχος 2011 Ντόρφμαν και άλλοι ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίσατε όλοι αυτό δεν μπορεί παρά να είναι θετικό 2011 λοιπόν Μισό λεπτό λέει ο πρόεδρος. κάνουμε κι άλλο άλμα. 2055 downtown υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2056 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2056 downtown ηλεκτρονικός έλεγχος για την 2056 ψηφίσατε όλοι Απορρίπτεται. 2053 ταραμπέλα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2010. Κατά. Απορρίπτεται. 2058 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2059 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2060 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2061 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2062 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2063 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2064 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 2065 υπέρ, κατά, έλεγχος. 2065 Σιλβέστρης, ηλεκτρονικός έλεγχος που ξεκινάει. 2065 απορρίπτεται. 2066 υπέρ, 2066 Καταρίνα Νεβεντάλοβα αντίθετη απορρίπτεται. MV32 μετά, υπέρ της MV32, κατά, απορρίπτεται. 2068 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2069 υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. 2070 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 95 του συγητού υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2073. Α, μισό λεπτό. 2073 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 96 του συγκητή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2074 Χάουσλινγκ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται μάλλον. 2075 Νταντέν υπέρ, κατά, έλεγχος, απορρίπτεται. Έλεγχος για την 2075 Νταντέν σας παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη. 2075 έλεγχος στα γρήγορα, πέρας ψηφοφορία. απορρίπτεται. 2076 περ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2077 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 2078 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 97 του συγκητού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2079 Λεγιάρικ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εγκρίνεται λέει ο πρόεδρος. Εγκρίνεται. 2080 Άλβες υπέρ κατά απορρίπτεται μάλλον 2082 υπέρ κατά απορρίπτεται θέλετε να γίνει έλεγχος όχι 2082 έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία για την 2082 Κάσια Περές και άλλοι ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται 2083 2083. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 2084 υπέρ, 2084 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άρθρο 39, 2085 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2086 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος, έλεγχος, 2086 έλεγχος. Έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. 2096. Πρέπει να ψηφίσουμε την 2094. 2094 λοιπόν, Νίκολσον, υπέρ. Υπέρ, κατά. Δεν βλέπω. 2094 παρακαλώ έλεγχος. 2094 Νίκολσον. 2094. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Απορρίπτεται. 2096 Νταντέν. Υπέρ. 2096. Υπέρ όλοι. Κατά εγκρίνεται. 2097. Σμιτ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται μάλλον. Ή... Μισό λεπτό. Ένα αλματάκι. 21-26 Σμιτ. 21-26 υπέρ. 21-26 υπέρ κατά απορρίπτεται έλεγχος 21-26 ηλεκτρονικός έλεγχος Σμιτ άρχεται η ψηφοφορία εγκρίνεται 2141 υπέρ. 2141 Λεγιάρικ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ. 99 κατά. Απορρίπτεται. 2144 Καλινόφσκι υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται μάλλον. Έλεγχος για την 2144 Καλινόσκη. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ισοψηφία. Συνεπώς απορρίπτεται. 2145. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2148. Έλεγχος. Καλώς. 21.45 Νίκολσον. Έλεγχος. 21.45. Ψηφίσατε όλοι την 21.45. 21-21 απορρίπτεται. Παρατρίχα. Καλύτερη τύχη την επόμενη φορά. 21-48 Dodge. 21 2148 κατά υπέρ κατά απορρίπτεται. 2150 υπέρ κατά απορρίπτεται. 100 του συγκητού υπέρ κατά απορρίπτεται. 2152 λεγιάρικ υπέρ κατά απορρίπτεται. 2153 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 2154 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 2155 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2156 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στο άρθρο 40. 2157 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 2158 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 2160 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 2161 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 2159 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 41. 2162 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 2163 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2164, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2165, 2166, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2167, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2167, 2168, υπέρ, 2168 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο. Όχι, 2169 υπέρ, 2169 Νίκολσον, κατά, απορρίπτεται. 2170 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2171 Ντελάουνς υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2173 τρεμόζα κατά απορρίπτεται 2172 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2170 α δεν είναι 2177 Στάρντι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2178 Στέρντι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2179 χαουσλινγκ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. MV33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2180 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 2182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2183 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2185 Dodge υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2186 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2188 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2187 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άλλο μικρό αλματάκι. Άρθρο 2276 τροπολογία Μάγερ υπέρ 2276 2276 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Διευκρινίστε τον αριθμό παρακαλώ Πρόεδρε 2276 υπέρ κατά εγκρίνεται 2277 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Θέλετε έλεγχο. Έλεγχος. 2277 Μάγερ. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Με μεγάλη διαφορά. 2278 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 10. Ρέτζι 10 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2279 Μάιερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2280 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2281 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 μισό λεπτό 2284 Μάιερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2285 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος έλεγχος μάλιστα ευχαριστώ δεύε 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20... 108 του εισηγητού 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Να περάσουμε τώρα στα εκτιμώντες. Είναι λίγα, λίγα και κατόπιν θα κάνουμε διάλειμμα. Να ξεκινήσουμε με το εκτιμώντα 112 μαγκίνες, υπέρ. Λουίς, 112. Υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Όχι να ελέγξουμε. Ελέγχουμε το εκτιμώντας 112. Πέρας. Απορρίπτεται για μία ψήφο. 113 πατράων έβες. Περ. Μετά. Εποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Budget 1. Όχι. Κοντ 1. Υπέρ κατά που εγκρίνεται. Dev 1. Υπέρ. Μπορούμε να ελέγξουμε το κοντ 1. Κοντ 1 γιατί το εκτιμώντα ένα αλφα ναι. Μάλιστα, να ελέγξουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Για να είμαστε σίγουροι. Κόντα 9. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ένα λεπτό. Ψηφίστε. Ψήφισε. Ψήφισατε όλοι. Θα καλό είναι ένα, ναι, αλλά δεν ψήφισε. Εγκρίνεται. Μάλιστα. Δεβένα. Υπέρ. Κατά. Το λίγο ότι απορρίπτεται. Πάμε. Κοντ 2. Περ. Κατά. Οχές. Εγκρίνεται. Κοντ 2. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφορία. Ψηφίσα Ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται. 117. Κάντεμπαχ. Δεν υπάρχει ψηφορία γιατί θετήθηκε η Ντεβένα. Όχι, δεν υιοθετήθηκε. Απορρίπτεται. Πρέπει να ψηφίσουμε. Μάλιστα, μάλιστα. 117 πρέπει να ψηφίσουμε. Υπέρ. Γιατί απορρίφθηκε η Ντεβένα. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Κον 3 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 127. Δεξιά υπέρ, και λυπή υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. ένα του συγκριτή Κον 4 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται θα έλεγα. Και τώρα περάσουμε στην τροπολογία Μαρινέσκου 165 υπέρ, κατά εγκρίνεται 167 τα μπάτζι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 συγητής υπέρ, κατά αποχές απορρίπτω. άλμπα ακόμη. Πάμε στροπολογίες κατά 2,70. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Κοντρόλ 7. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 279 λίγο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα. 312 Παύλο Άλβες υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται 313 Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 314 υπέρ Κατά εποχές εγκρίνεται 3.11 όχι 3.15 3.15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 324 Στίβενσον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Λοιπόν, δύο τελευταίες ψηφοφορίες, προσοχή. Θα ψηφίσουμε την πρόταση για την απόφαση να διάλεξη για πραγματική ολίδη οργανική βάση του άρθρου 70-270α υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφορία. Συγγνώμη. Άρχεται η ψηφορία. Ψηφίστε το όλοι. Για το ΕΛΚ υπάρχει μία ψήφος παραπάνω. Ψήφισατε όλοι. Μάλιστα. Εγκρίνεται. Και τώρα απόφαση για τη διαπραγματευτική ομάδα που θα αποτελείται από τον πρόεδρο, τον συζητητή και τους κοιόδης. Άρχεται ψηφοφορία υπέρ. Ηλεκτρονικά. Κατά. Και εγκρίνεται με ευρία πλειοψηφία. Ευχαριστούμε. Κάναμε το πρώτο βήμα. Σας ευχαριστώ όλους. Κολέγοι, 15 minuti. 15 λεπτά διάλειμμα, συνάδελφοι. 15 λεπτά και ξεκινάμε από τώρα. Iniziamo. Να ξεκινήσουμε παρακαλώ. Bene. Innanzitutto ευχαριστήσω τον Λουίς Κάπολα που είναι εισηγητής και φυσικά και όλους τους σκιώδεις εισηγητές. Κάναμε ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Να περάσουμε τώρα στην αγροτική ανάπτυξη. Θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή συνεδρίαση σήμερα το πρωί με την αγροτική ανάπτυξη και το απόγευμα θα ψηφίσουμε την ενιακόα. Και φτάνει τη χρηματοδότηση της κοινή γερικής πολιτικής ε, θα την ψηφίσουμε αύριο το πρωί. Εντάξει. Συνεχίζουμε με τους ίδιους κανόνες και εδώ έχουμε ένα κατάλογο ψηφοφοριών που ακολουθεί τις 37 συμβαστικές τεχνολογίες. που θα ψηφιστούν σε μπλοκ για μια ακόμη φορά. Λουίς, να σου δώσω το λόγο, το θες, όχι. Λοιπόν, να περάσουμε τότε στην ψηφοφορία. Είστε έτοιμοι? Περνάω στο άρθρο 74, με συγχωρείτε, Ρέιμερ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσα το όλοι. Αέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 του συγητή. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Όχι, τα χειρός, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11, Ρέτζι υπέρ. Κατά, εποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 12, Ρέτζι υπέρ. Κατά, εποχές, απορρίπτεται. 13, Ρέτζι υπέρ. Κατά, εποχές, απορρίπτεται. 14, Ρέτζι υπέρ αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 14 Ranger έρχεται ψηφορία αέρας εγκρίνεται Ε, Προσοχή. Φαίνεται να έχουμε δύο ψήφους παραπάνω ποιος μπορεί να ψηφίσει και ποιος δεν μπορεί. Υπήρχε πάντως η πλειοψηφία, προχωρούμε. Δεν 209 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 7 εισηγητής υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 15 ρέτζι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 211 άλβες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 212 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 213 υπέρ. Συγγνώμη, 2.15 υπέρ κατά εποχές θα έλεγα απορρίπτεται 2.16 2.18 2.18 Σάρμπου. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.19 Δαντάν. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.20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 κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Έλεγχος το 29. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Και πάλι έχουμε μία παραπάνω ψήφο. Υπάρχει ένας παραπάνω που ψηφίζει. Ο κύριος Ανιώ, παρακαλώ. Πρόεδρε, αυτό δεν είναι ικανοποιητικό. Έχουμε μερικές φορές ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία και βλέπουμε ότι ψηφίζουν παραπάνω και κατόπιν συνεχίζουμε με την άρθρηση χειρός ε, και μπορεί να συνεχίσετε το λάθος, μπορούμε πώς να το επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα τώρα. Μάλιστα να προχωρήσουμε πιο αργά για να μην έχουμε μπερδέματα. «231. Λαβία. Υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 2.32 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 4 κόντ υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 2.33 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 16 Ρέτζι. Πάμε στη 239 Λαβία. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.40 υπέρ. Κατά. Αποχές Γκρίνεται θα έλεγα. Θέλετε να κάνουμε έλεγχο. Σαντζε Σμιτ. Άρχεται η ψηφοφορία. Σωστό τώρα. Εγκρίνεται. 2.41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτει. 2.42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτει. Για το 2.42 θέλετε έλεγχο, μάλιστα. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. 2.42. Εγκρίνεται. κ. τον Γκάμπριελ, υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 2.49. Υπέρ. Κατά. εποχέ Απορρίπτεται. 2.50. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 2.52. Υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 2.54 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 2.55 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 2.56 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 256 σκοτά και λυπή. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 257 υπέρ. Κατά. Αποχές θα έλεγα απορρίπτεται. 258 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 259 υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 260 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 261 υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 262 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 264 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 265 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 267 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 268 υπέρ. Κατά αποχές. Λοιπόν, να ελέγξουμε το 268. Αερά συγκρίνεται. Αυτρία Ρέτζ 17 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 269 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 270 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 273 πατράων έβες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 274 ταραμπέλα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το 75 Ρούμπιξ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το 76 Per. κατά αποχές απορρίπτεται. Το 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, συγγνώμη, 2, 78 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 του συγητή. Υπέρ. Κατά, Αποχές εγκρίνεται. Τώρα, να μπούμε στους συμβιβασμούς. Συμβιβασμός 1, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Συμβιβασμός 1, εγκρίνεται. Συμβασμός 2. Ηλεκτρονική ψηφορία πάντα για τους συμβασμούς. Άρχη ψηφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. NV32. Δεν χρειάζεται ηλεκτρονικά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος NV32. Άρχεται ψηφορίας. άρθρο 6, 32. Σβήσετε όλοι. Εγκρίνεται. Να ξαναπροσπαθήσουμε. MP32. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε όλοι. Εγκρίνεται. 6 Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Συμβασμό 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Περνάμε στο συνδεσμό 4 ηλεκτρονική ψηφορία. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 484 Δανέλης. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ελεγχώ. 484 Δανέλης. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. NV35 υπέρ. υπέρ. Άρθρο 9. Κατά. Απορρίπτεται. έλβη LV35. Εντάξει, πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε στο ε, Κάντιμπαχ 561 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 562 Σμιτ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. NV36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 563 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. 564 υπέρ. Κατά. εποχές απορρίπτεται. 566 σμίτ υπέρ. Κατά. εποχές απορρίπτεται. Έλεγχος 566 σμίτ. Ψηφίστε. Πέρας. Απορρίπτεται. MV37 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 569 φέρμ και λοιπή. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 570 φάιμον. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 571 υπέρ κατά Εποχές απορρίπτεται. 572 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 574 δαντέν, υπέρ. Κατά. εποχές να κάνουμε έναν έλεγχο για το 574-75. Έρχεται η ψηφορία. Αέρασε. Απορρίπτεται. 575 σμίτη υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 576 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 577 γουτιέρε και λοιπή υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται 578 υπέρ συγγνώμη Ρέτζι 34 υπέρ κατά Αποχέ απορρίπτεται Ρέτζι 35 υπέρ κατά αποχές Να ελέγξουμε, έρχεται ψηφορία. 35 ρέτσι. Εγκρίνεται. Πέντε υπέρ. Κατά, εποχές, εγκρίνεται. 584 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 της υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Φαϊμό 585 υπέρ κατά απορρίπτεται 37 Ρέτζι υπέρ κατά αποχές 1.38 NV38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 πόντ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 588 σάρμπου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 38 ρέτζι υπέρ κατά απορρίπτεται. 589 μπας υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 40 ένβη υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 590 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 592 Dorfman υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτω. 593 υπέρ. Κατά. Αποχές. Γκρίνεται θα έλεγα. Να ελέγξουμε την 593 Ντόρφμαν. Αρχή. Ψήφισατε όλοι. Απορρίπτεται. 594 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 595 Ντόρφμαν υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 596 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 11, 605 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται θα έλεγα. 606 Μάιερ υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 607 Νίκολσον υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 609 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 612. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 614 γουτιέρες υπέρ. Κατά. Οχές. Εγκρίνεται. 616 υπέρ. Όχι. Συγγνώμη, 618. Μάιερ υπέρ. Κατά. Πεχές εγκρίνεται. Ξεκούσα 18. Να το δούμε. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε. Ψηφιστόλη. Απορρίπτεται. 619 Νίκολσον. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 621 υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 625 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 629 υπέρ κατά εγκρίνεται 632 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται Να πάμε στο 633 Μάιερ υπέρ. Υπέρ κατά. Εγκρίνεται. 634 Χάρκιν υπέρ. Κατά αποχές υπορρίπτεται. Τώρα, 6.36 σκοτάκι λυπή υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 6.37 υπέρ, όχι. 6.38 Γκουτιέρες, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 11 κοντ, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. 11 κοντ. Αρχή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρασε. Απορρίπτεται. Πολύ ωραία. Συμβεσμός 5, ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ευραίος. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το συμβασμό 6, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο συνδεσμό 7. Άρχεται η ψηφορία του συνδεσμού 7. Ψήφισε όλοι. Ποιος λείπει. Ελέγξτε να έχει ανάψει το λαμπάκι. Εγκρίνεται ο συμβιβασμός αυτό. Συμβιβασμός... 8. Άλλο ένα άλμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Λοιπόν, ψηφίσατε όλοι. Για το 8. Ευρία πλειοψηφία υπέρ. Πρέπει να ψηφίσουμε. NV59. Άρθρο 19. Υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 907 σμιτ. Υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. 908, δηλαδή υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. 909 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 910 Λιγέρικ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 911 σκοτά και λίπε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9-12, Νταντάν, υπέρ. Κατά αποχέ απορρίπτεται. Τώρα, ηλεκτρονική ψηφοφορία για το συμβιβασμό 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνει. Ακόμη ένα άλμα και πάμε στο συνδεσμό 10. Άρχεται η ψηφορία για το 10. Πέρας. Εγκρίνεται. Άλλο ένα άλμα. Πάμε στο 21. 1083 Κάντεμπαχ. Υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. Χίλια υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα πάμε στα μπλοκ. Έχουμε ψηφορία σε μπλοκ, συμβιβασμός 11 με ηλεκτρονική ψηφορία. και 15 έρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Μόνο μία ψήφο κατά είχαμε. Περνάμε στο 1089. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Facciamo un altro salto. Κάνουμε κι άλλο άλμα. Andiamo al compromesso 16. Συμβαστική 16. Συμβαστική 16. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Καλώς και εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. Άρθρο 29. Block vote, επιλογή Β. Ηλεκτρονικά. Άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Attenzione, blocco voto Ομάδα ψηφοφοριών επιλογή Β, option B. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πάμε στην άλλη ομάδα, επιλογή Α. Πάντα με ονομαστική ψηφοφορία, option Α. Ε, ξεκινάει ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για την option α, την επιλογή α, πέρας. Απορρίπτεται. Δεν ψηφίστηκαν οι δύο αυτές ομάδες τα δύο μπλοκ, πρέπει να ψηφίσουμε τις τροπολογίες μία-μία. Μόνο τέσσερις σελίδες. Ξεκινάμε. 1289 Σμίτ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1290 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1291 Γέγκλε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται μάλλον. Έλεγχος της 12.91 Γέγλε. Ηλεκτρονικός έλεγχος. 12.91. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 12.92 Σμιτ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12.93 Ντελάνζ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται μάλλον. Πρέπει να κάνουμε έλεγχο. να σηκώνετε καλά τα χέρια για να πηγαίνουν πιο γρήγορα. 1293 αντελάμους ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. 1293. Εγκρίνεται. 12.94 υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51 Ρέτζι. Όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. 7 Ντεβε υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12.97 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1298 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1299 υπέρ όχι Θέλετε να κάνουμε έλεγχο για τη 1298 Κόστιγκερ. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 1298 Κόστιγκερ. Ψηφίσατε όλοι 1298 εγκρίνεται. «1305 φαϊμών». «1305 υπέρ» κατά αποχές απορρίπτεται. «1306 υπέρ» κατά αποχές απορρίπτεται. «1307 υπέρ» κατά αποχές απορρίπτεται. 1308 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 1309 υπέρ, κα, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1310 ράιμερς υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 1311 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 1313 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 1312 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 1314 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 96 ένβη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1315 χάρκιν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1316 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1317 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1318 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1000... Θα κάνουμε έλεγχο. 1318 δες έλεγχος. Έλεγχος για τη 13-18 δες Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται 1318. 1323 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 του συγκητού υπέρ. 42 υπέρ. Κατά. Μάλλον απορρίπτεται. 1324 ροντ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1325 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1326 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1327 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1328 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1329 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1330 Σμιτ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1331 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Un momento, eh. 37. Sì. 13-37. 13-37 ταραμπέλα iper. Υπέρ απορρίπτεται. 1338 Κάντεμπαχ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο, γιατί. Γιατί 1338. Για τη 1338 ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. 1338 Κάντεμπαχ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε στη 1340 Σμιθ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 1340 Σμιθ υπέρ, σηκώντε καλά τα χέρια παρακαλώ, 1340 Σμιτ υπέρ, κατά, καλώς απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την NV98 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 1341 ράιμερ υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 1341 έλεγχο Άρχεται η ψηφοφορία Γιατί τη 1341 Ρέιμερ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 1342. Α, 1343. 1343 Κάντενμπαχ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1344 Κάντενμπαχ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στις συμβαστικές. Συμβαστική 19 με ηλεκτρονική ψηφοφορία που άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με τις συμβιβαστικές. Συμβιβαστική 20. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβιβαστική 20. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται η συμβιβαστική 20. Συνεχίζουμε. Ψηφίζουμε μαζί τη συμβαστική 21-22, 34 και λοιπά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνονται. Κάνουμε κάποια άλματα. Πολύ καλά. Άρθρο 34. 1460 Σμίθιπερ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεκατέσσερα εξιντένα Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την 1462. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1463 Σμιτ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 48 του εισηγητού υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1464 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1465 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 1466 Πόλσαν και άλλοι υπέρ, κατά 1466 έλεγχος παρακαλώ. 1466 ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συνεχίζουμε λοιπόν. 1467 ρόντου υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 1468 φεϊμών υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 1469 Εράνς Γκαρσία και άλλοι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 1470 1471 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1472 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Δεκατέσσερα υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. Δεκατέσσερα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 1475 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1477 ρέιμερς, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1477 έλεγχος έλεγχος για τη 1477 Ψηφίσατε όλοι. Για 1477. Πέρας. Εγκρίνεται. 1481 ογδόντα Κάντενμπαχ υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1482 ρόντους υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 1483 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 1484 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Πάμε στην βεστική 23. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη συμβιβαστική 23. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την ΔΕΒΕ 8. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην ΔΕΒΕ 9. ΔΕΒΕ 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία ψηφίζουμε τώρα τη συμβιβαστική 24. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίστε καλά παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Τη συμβαστική 24 που εγκρίνεται. Συμβαστική 25. Συμβαστική 25 με ηλεκτρονική ψηφοφορία η οποία ξεκινάει. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 26. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη συμβαστική 26. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έχουμε κάποιες ψηφοφορίες. Τροπολογία 59 του συγκητού υπέρ. Διανατάσσεις της χειρός. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16-16 Ντόρφμαν, πρώτο τμήμα υπέρ. Σηκώστε το χέρι παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 27 ηλεκτρονική ψηφοφορία που ξεκινάει. Συμβιβαστική 27. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το 41, 1665, Ρόντους και Άλτρι. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έχουμε κάποιες ψηφοφορίες τώρα. 1667 Μάγερ. υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. 1668 Πόλσεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 42, 1670 Σικιέρσκι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1671 Γκουτιέρες υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τώρα 1672 Σικέρες και υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μάλλον. Όχι. Έλεγχος. Για τη 1672 ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίστε, ψηφίστε. 1672 έλεγχος ηλεκτρονικός. 1672 σε Κυρέσκι. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται λοιπόν. Διανατάσσω στις χειρός τώρα. 1673 υπέρ. 1673 Πρέντεργαστ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 1674 Κάντεμπαχ υπέρ κατά δεν θα λέγω 124 όχι όχι όχι όχι ΕΝΒ. 64 Ρέτζι υπέρ κατά απορρίπτονται. 123 ΕΝΒ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στο άθρο 44 της ΔΕΒΕ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1676 Σικέρσκι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1677 Κουτιέρες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 δεύε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1678 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1679 καρόνα υπέρ. Α, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. «1680 υπέρ» Κατά. Έλεγχος. Νομίζω ότι είναι υπέρ. 1680. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άλαμπαρτ και άλλοι. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Να δούμε αν εγκρίνεται ή αν απορρίπτεται. Α, απορρίπτεται. 1681 Νίκολσον στο άρθρο 45. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16, 83, Γκουτιέρες και άλλοι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πάμε τώρα στις συμβιβαστικές με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Συμβιβαστική 28 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. Άρθρο 49, 17-26, κουτιέρες υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 17-27 ταραμπέλα υπέρ. Υπέρ, κατά, κατά, αποχές απορρίπτεται. 17-28 γέγλε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται μάλλον. Έλεγχος για τη 17-28 γέγλε. 17-28. Μάλλον εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 17-29 σκοτά και άλλοι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 17-30 κάντεμπαχ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 17-31 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 17-32 γιάρ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 17.33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17.42 φεϊμού υπέρ κατά απορρίπτεται. 1743 Γκάμπριελ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1744 Τεραμπέλα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1745 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1746 Μάιερ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1748 γιάρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1750 φεϊμού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1751 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 17.55 φεϊμού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17.56 φεϊμού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17.57 και υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17.58 φεϊμού υπέρ κατά άποχες δεν ξέρω 1758 έλεγχο σας παρακαλώ 1758 μου. πέρας εγκρίνεται εγκρίνεται Πάμε στην 1760. Φεϊμό υπέρ 1760. 1760 φεϊμών υπέρ κατά εγκρίνεται 1761 1761 φεϊμόν υπέρ κατά απορρίπτεται αυτή τη φορά 1762 Κόστιντζερ υπέρ κατά εγκρίνεται 1763. Σμιτ, θέλετε να κάνουμε έλεγχο. Συγγνώμη, έλεγχο για τη 1762 Κόστιντζερ. Άρχεται την ψηφορία 1762. Εγκρίνεται 17, 63 σμιτ, υπέρ. Κατά, εποχές, εγκρίνεται. 1764 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1765 Κόστιγκερ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1767 Φαϊμόν υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 1768 Μάιερ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1770 Γκουτιέρης και λοιπή υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να κάνετε έλεγχο, όχι. Ε, μάλιστα, έλεγχο 17.70 70 γιατί μου το ζητάει αντιπρόεδρο, δεν μπορώ να αρνηθώ. το όλοι. Απορρίπτεται. Φεϊμούν 1775 υπέρ παρακαλώ μανατας χειρός κατά απορρίπτεται 1776 υπέρ κατά απορρίπτεται 1777 υπέρ κατά απορρίπτεται 1778 Μάιερ υπέρ κατά εγκρίνεται 130 NV υπέρ κατά εγκρίνεται. 1779 Γκάμπριλ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1781 Νταντέν υπέρ κατά αποχές αλλά ναι, αλλά κάνουμε ένα έλεγχο για την τροπολογία Νταντέν 1781. Σβήσατε όλοι. Πέρας. Υπέρ. Λοιπόν, το 1783. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 1784. Φαϊμό. Όχι. 86. Άντσιλα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται λέει υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 1787. 88 με συγχωρείτε υπέρ. Εποχές εγκρίνεται. 1789. Υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 1791. Πόλσεν υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 1792 Γκάμπριλ, υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 1793 Μάιερ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 1794 Καντέκ υπέρ. Κατά. εποχές, απορρίπτεται. questo blocco. Andiamo a fare un voto. Να περάσουμε σε ηλεκτρονική ψηφορία για το συνδεσμό 29α, 29β και 30 του CGT. Άρχεται ψηφορία. Ψηφορία σε μπλοκ. 29α, 29β και 30. Άρθρο 61 έως 63. το όλοι. σε ευρία πλειοψηφία. ΔΕΒΕ 12. Ανάταση χειρός, υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 13. Ανάταση χειρός. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. με ηλεκτρονική ψηφορία να πάμε στην ε, τροπολογία 31-33, άρθρο 64, αρχή ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Αέρος. Εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε τώρα τη 1963 Γκάμπριελ. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Έλεγχος παρακαλώ. 1963. Έχω το ψηφορία για έλεγχο. Πέρασε. Πάμε στο άρθρο 66. Μενάτας χειρός 19, 89, 1990 υπέρ, κατά, γκρίντ. Άρθρο 67, 1999, πατρόν έβαση υπέρ. κατά εποχές συγκρίνεται. Δύο χιλιάδες σκοπά και λίγο υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2001 Αλαμπάρτ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2002. Τραμός υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2003. Λαβία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2004 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συνεχίζουμε. 2005. Δόρφημαν. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2006 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 κόντ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20.07 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Δείτε 9 καντέκ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2010, Κόστιγκερ, υπέρ, κατά. Δεν μπορείς να είσαι κατά, είναι δική σου η τροπολογία. Λοιπόν, επαναλάβουμε. 20-10 Κόστιντζερ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Έλεγχος. Είναι ευρία πλειοψηφία, αλλά ας αλλάξουμε την 2010. Πέρυσι. Εγκρίνεται. 12, 2012, δώδεκα, Ντόρφμαν. πίπτη, συγγνώμη με Κάντεμπαχ υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 2019 Γκουτιέρες υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 22 Μάιερ υπέρ αυτά. απορρίπτεται 70 εισηγητή υπέρ κατά έλεγχος για το 70 άρχεται η ψηφορία πέρας και απορρίπτεται 20-23 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 20 κόντ υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 20-24 εγκλη υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 20-25 σκάντελμος υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 20-26 υπέρ, κατά, εποχές απορρίπτεται. 20-27 πατρονέδες υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 20-28 κάντεμπατ υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 20-29 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 75 Ρέτζι. Υπέρ. Αυτά αποχές απορρίπτεται. 20-30 υπέρ. κατα αποχε αποχές απορρίπτεται. 20-31 Κάντελμπαχ υπέρ. Κατά αποχε απορριπτεται απορρίπτεται. 20-32 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτω. 233 και σκυπέρ κατά Εποχέ. εγκρίνεται 2034 υπέρ κατά Εποχέ. απορρίπτεται 2035 υπέρ κατά απορρίπτεται άρθρο 82 236 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Είκος τριντεφτά Ντόρφμαν υπέρ. Κατά. He wants a check in 2036. Yes. Okay. Uh, è stato chiesto un controllo. Ζητήθηκε έλεγχος ψηφορίας για την 2036. Άρχεται η ψηφορία. 2036. Ψηφίσατε όλοι πέρασε. Δεν Είκοσι σαράντα ένα μάγερ υπέρ. Απορρίπτεται. 78 ρέτζι περ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20-42 φημών πέρ, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Gutierrez Per Κατά. Αποχές Πόσο 244 άντρου υπέρ. Κατά. Αποχές Μήπω 245 ράντ υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 246 μπεραντίκ. Όχι. Γέκλο. 247 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 2052 υπέρ κατά απορρίπτεται 2053 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 2056 δόρφμαν, υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 57 αντιλάζ υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. 258 και υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. Μάιερ 259 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 260. 21 κοντ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι. Ελεγχο. Για την 21 κόντ. Απορρίπτεται, έχετε δίκιο. 20-62 Πόλσεν. Υπέρ. Με να τα σχηρώσω. Κατά εποχές απορρίπτεται. Είκοσι έξι Υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 67, εφτά, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Πάμε στην 269. Υπέρ, κατά, 2070, Παστάμκο, υπερ υπέρ. Κατά. 2071, Ροντ. Υπέρ. Κατά. 2072 υπέρ κατά απορρίπτεται 2076 Φρανσίσκο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται με ένα χειρός 139 ένδυ υπέρ κατά εγκρίνεται σωστά να ελέγξουμε για την 139 NV παρακαλώ. Ψήφισατε όλοι. Εγκρίνεται. Είκοσι εβδομήντα εφτά Κάντερμπαχ, υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. Άρκιν 2081 ε, περ κατά εποχές εγκρίνεται 20 84 Παμπεστάμκους υπέρ κατά εγκρίνεται 2085 Αλαμπάτ υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 140 ένβη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 288. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 290 ρόντους. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 291. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Να κάνουμε έλεγχο για την 2091 Μπεραντίκ. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 2093. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 295 κατά αποχές απορρίπτεται. 294 άλβες κατά αποχές απορρίπτεται. 296 πέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. 298 πέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2106 Ράιμερς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 21.07 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Όχι. Συγγνώμη. 21.07 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 21.08 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Έλεγχος. Μάλιστα. Για το 21.08. Γκουλάρ. Εγώ θα λέγω ότι εγκρίνεται, αλλά για να δούμε. Όχι, απορρίπτεται. Μάλιστα. 21.09. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 21.11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21.12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21.13. Όχι. άλμα. 21-22 νταντά. Υπέρ. 21-22. Υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 145 ένβη. Υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. Πάμε στα εκτιμώντας. Ένα ντεβε υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. Ένα κοντ υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. Ένα ρέτζι υπέρ. Κανείς. Υπέρ. Κατά. Μάλιστα, απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 83 λαβή και λυπή. Υπέρ. Κατά. Θα έλεγα γκρίνεται. Να κάνουμε έλεγχο. Για την 83. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται. NV2 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 3 NV υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 96 Μπεραντίκα υπέρ κατά θα έλεγα απορρίπτεται 98 Πατρέων υπέρ κατά εγκρίνεται 99 υπέρ κατά εγκρίνεται

7 envy, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 5 reds, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ένα λεπτό, νομίζω πρέπει να είμαστε στο συμβασμό. Ένα λεπτό. Σχεδόν τελειώσαμε. Sì, sì. Eh. Sì, sì, sì, sì. 174. 174 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 2, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα 184 πρεντεργαστή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 187 μπαραντίκα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 190 παρα 190 υπέρ κατά εποχέ απορρίπτεται Ρέτζι 9 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 196 Βέστλουντ και λοιπή υπέρ κατά απορρίπτεται 202 Πόλσεν υπέρ. Κατά. Έλεγχος. 202 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται. Ρέτζι 10 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Ηλεκτρονική ψηφορία υπέρ. Πέρας. Απορρίπτεται. Δύο τελευταίες ψηφοφορίες ηλεκτρονικές. Άρχεται Και ψηφοφορία για την πρόταση και για να ξεκινήσουν οι διοργανικές διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τους κανόνες του 72 και του 70α. Άρχεται ψηφορία. Πέρασε. Ευρεία ψηφία, υπέρ. Τελευταία ψηφοφορία για τη διαπραγματευτική ομάδα όπως για τις άμεσες ενισχύσεις από τον πρόεδρο, τον συγγητή και του Σκιώδης. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώσαμε και την ψηφορία για την αγροτική ανάπτυξη. Συγχαρητήρια στον κύριο εισηγητή, στον κύριο Καπούλα Και συγχαρητήρια και σε όλους τους κοιόδης εισηγητές. Θα συνεχίσουμε την ψηφοφορία το απόγευμα για την ενιαία ΚΟΑ του κ. Νταντέν στις 3. Αλλά ένα λεπτό, ο κύριος Ολένιτσακ ζήτησε το λόγο. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja mam pytanie, czy nie moglibyśmy przesunąć e, jutrzejszego głosowania. Έχω την εξή ερώτηση, Πρόεδρε. Μπορούμε να μετακινήσουμε την ψηφορία που έπρεπε να λάβει η χώρα αύριο και να την κάνουμε σήμερα την αυριανή ψηφοφορία, πώ θα μπορούσαμε να την κάνουμε σήμερα, φαίνεται ότι έχουμε αρκετό χρόνο να ολοκληρώσουμε σήμερα τι ψηφοφορίε. Είναι το τέταρτο, ο τέταρτος φάκελος, εξηγητής ο κ. Λαβία, αύριο θα ψηφίσουμε, γιατί σήμερα ο εισηγητής ε, έχει ζητήσει να μην γίνει αυτή η ψηφορία. Θα ψηφίσουμε μόνο την έκθεση Νταντέν σήμερα το απόγευμα. La parola Giovanni Lavia. Giovanni Αν συμφωνεί ο κ. Λαβία, εγώ πιστεύω, Παόλο, ότι δεν είναι ένα θέμα αιτήματο του συγητή. Απλώ πρέπει να δούμε αν όλοι είναι διαθέσιμοι να συνεχίσουν την ψηφοφορία απόψε. Επειδή θα είμαστε κουρασμένοι από την πλευρά τη δική μου, δεν υπάρχουν προβλήματα ως εισηγητής. Πρόεδρος, ένα λεπτό, συνάδελφοι, προσοχή, ένα λεπτό. Λοιπόν, ε, έχουμε τον κανονισμό της νέας ΚΟΑ, αν πάει καλά η ψηφοφορία, όπως σήμερα το πρωί, εγώ θα πρότεινα να κλείσουμε απόψε και με τη χρηματοδότηση της ΚΑΠ. Αν όμως αντίθετα υπάρχουν δυσκολίες, τότε θα ψηφίσουμε αύριο. Υπάρχουν αντιρρήσεις? Ωραία. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή σας όρεξη. Θα ξαναπούμε στις 3.